Uh, Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας συνεχίσουμε την εργασία μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πασκάλ Λαμή, Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και την κυρία Βάλεντιν Ζουμπορίσκα, αναπληρώτρια, Γενική Διευθύντρια. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν για σας να φτάσετε στις Βρυξέλλες. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς η ευκαιρία που έχουμε να σας υποδεχθούμε εδώ στην Επιτροπή μας μετά τις συναντήσεις που είχε με εσάς η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γενέβη στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου επί τη ευκαιρία της τελευταίας Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας υποδεχόμαστε κύριε Λαμή εδώ διότι ως αρμόδιος επίτροπος για το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπιστήκατε ενεργά τον ρόλο του Κοινοβουλίου και τη συμμετοχή τους στη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Έχετε συμμετάσχει επίσης ε, στη σύνταξη της νέας συνταγματικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αρχίσει πλέον να ισχύει, έχει τεθεί σε ισχύ πιστεύω ότι ίσως οφείλουμε πολλά, διότι στηρίξατε την ανάδειξη και την αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει ριζικά η κοινή εμπορική πολιτική, ειδικότερα όσον αφορά στους ενισχυμένους πυλώνες που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή και την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενισχύεται λοιπόν το προφίλ του Κοινοβουλίου που είναι και το θεσμικό όργανο το οποίο είναι το μοναδικό που εκλέγεται άμεσα από τους λαούς της Ευρώπης. Έχουμε συνεργασία με εσάς, αλλά και με τον οργανισμό που εκπροσωπείτε και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις προτάσεις σας για το πώς το Κοινοβούλιο μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις νέες δυνατότητες που του έχουν δοθεί. Βεβαίως θα μάθουμε και πολλά για την κατάσταση που επικρατεί ως προς τις διαπραγματεύσεις για το γύρο της Ντόχα. Στην τελευταία υπουργική διάσκεψη στη Γενέβη είχαμε την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τα κράτη-μέλη πράγματι αναγνωρίζουν το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΟΕ στην απάλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τονίζεται η σημασία του ΠΟΕ και ως προς την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και ως προς την ευελτίωση των συνθηκών ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Άλλωστε, στο πρώτο τρίμηνο αυτής της χρονιάς θα γίνει η αξιολόγηση του κατά πόσο είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του γύρου, του γύρου της Ντόχα. Όλα αυτά θα φανούν πιο ξεκάθαρα στα τέλη Μαρτίου σε επίπεδο ανώτατων αξιωματούχων. Πολλοί επιθυμούν να δοθεί ε, μια λύση με βάση το πακέτο του Ιουλίου του 2008. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι βέβαια ακόμα έτοιμες να δεσμευθούν ως προς το πακέτο αυτό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει και υπουργική διάσκεψη πριν από το επόμενο G20, ώστε να καθοριστεί σε πολιτικό επίπεδο κατά πόσο είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του γύρου αυτού φέτος. Εσείς όμως ε, είστε εδώ για να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλωσορίσατε και πάλι κύριε Πασκαλαμή. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω και εγώ τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σε αυτή την αίθουσα και έχω την ευκαιρία να απευθύνω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλο που την τελευταία φορά που εμφανίστηκα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήμουν αντιμέτωπος με μια άλλη σύνθεση. Έχουμε τώρα νέα θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε νέα συνταγματική συνθήκη. Έχουν επέλθει λοιπόν σημαντικές αλλαγές από την τελευταία φορά που είχα έρθει εγώ εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις αλλαγές αυτές. Ο πρόεδρος της Επιτροπής σας αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα και έχει δίκιο. Πράγματι και εγώ έχω συμβάλει στη διατύπωση, στη σύνταξη, στη κατάρτιση αν θέλετε της ε, σημερινής συνθήκης της Λισαβόνας η οποία δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζουν μια εντελώς καινούρια θεσμική κατάσταση. Βρίσκεστε σε μια καινούρια θέση έχετε πολύ περισσότερες εξουσίες από ό,τι είχατε στο παρελθόν ως προς την ε, χάραξη των αποφάσεων αλλά και την παρακολούθηση των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με τη διεθνή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια έχετε και πολύ περισσότερες ευθύνες. Σίγουρα λοιπόν έχετε ένα πλεονέκτημα στη δουλειά σας, θα έχετε όμως και πολύ περισσότερη δουλειά να επομιστείτε και θα έχετε και πολύ περισσότερους συνομιλητές διαφόρων προελεύσεων. Και σίγουρα και στους κόλπους της κάθε πολιτικής ομάδας αλλά και εντός κάθε επιτροπής θα καλείστε να λαμβάνετε δύσκολες ενίοτε αποφάσεις διότι θα απαιτηθεί από εσάς να βρίσκετε συνενετικές ή συμβιβαστικές λύσεις σε αρκετά δύσκολα ζητήματα. Ε, μιλώ εντελώς ουδέτερα λέγοντας ότι με αυτές τις ε, καινούργιες αλλαγές θα ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή διαπραγμάτευση που διεξάγεται σε πολυμερές επίπεδο. Μια πιο ισχυρή ένωση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι εφικτή διότι έχει περισσότερη ισχύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι δηλαδή πιο δημοκρατική πλέον η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή όργανα και γι' αυτό θα έχει και περισσότερη ισχύ. Ως εισαγωγική παρατήρηση λοιπόν, επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να σας περιγράψω σε γενικές γραμμές το διεθνές σκηνικό περί του εμπορίου ώστε να περάσουμε στη συνέχεια σε πολύ πιο συγκεκριμένα ζητήματα προς συζήτηση. Αν δείτε το παρελθόν, σίγουρα θα γνωρίζετε ότι πριν από ένα χρόνο ήταν στο απόγειό της η κρίση παγκοσμίω. Είχαν καταρρεύσει οι εξαγωγές κατά μείον 40% οι εμπορικέ συναλλαγέ συρρυκνώνονταν δραματικά, η τραπεζική φερεγγιότητα ήταν εν κινδύνο και, το 90, και κατά 90% είχε μειωθεί ε, το, ε, οι εμπορικέ συναλλαγέ που ανέρχονται σε 63 εκατομμύρια παγκοσμίω. Αλλά και οι άμεσε ξένε επενδύσει είχαν μειωθεί ιδιαιτέρω. Υπήρχε μεγάλη ανησυχία ότι η κατάρρευση δηλαδή, του εξωτερικού εμπορίου θα οδηγούσε σε προστατευτισμό. Και ο προστατευτισμός, όπως γνωρίζετε, συνήθως κάνει την κατάσταση ακόμα, ακόμα πιο δύσκολη. Και γι' αυτό εμεί στο ΠΟΕ αμέσως προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε στενά τα διάφορα μέτρα ε, που είχαν να κάνουν με το εμπόριο, πάντοτε τηρώντας και εφαρμόζοντας τη βασική αρχή που πιστεύω ότι γνωρίζετε όλοι και η οποία είναι η εξής. Η διαφάνεια είναι και το καλύτερο απολυμαντικό. Βεβαίως υπήρχε και ανησυχία ότι λόγω της κρίσης οι δωρητές θα μείωναν την αναπτυξιακή βοήθεια και ήταν αυτό κάτι που μας απασχολούσε ιδιαιτέρως. Τα, κατά πόσο θα μειωθούν δηλαδή τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές. Η Βάλεντιν που κάθεται εξ αριστερών μου είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Την ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί σας, πολύ τη γνωρίζετε ίσως και θα αναφερθεί στο θέμα αυτό αργότερα. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν πέρυσι. Ένα χρόνο μετά, σήμερα δηλαδή, βλέπουμε μια ισχνή ανάκαμψη στις εμπορικές ροές. Στη σύνοδο G20 του Λονδίνου αναλήφθηκε δράση και έτσι αυξήθηκε η πιστοτική τα πιστοτικά μέσα που θα δίνονταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. οι δωρητές δεν αποσύρθηκαν από τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει, παρόλο που δεν έχουμε τα τελευταία στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία στη διάθεσή μας. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές όλοι έχουν αυτό περιοριστεί, αναφέρομαι κυρίως στις κυβερνήσεις και έχουν καταφέρει να κρατήσουν τις αγορές ανοιχτές. Βεβαίως δεν έχουμε ξεπεράσει το κίνδυνο. Αυξάνονται ενδεχομένως τα ποσοστά ανεργίας και οι οικονομίες συρρυκνούνται και όσο συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα ο κίνδυνος προστατευτισμού θα παραμένει. Επίσης, έχουμε ε, πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα πολυμερές σύστημα εμπορικών κανόνων κανόνες τους οποίους τηρούν οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν συγκεκριμένο κανονιστικό ε, πλαίσιο για την συμπεριφορά τους. Αυτό λοιπόν το πολυμερές εμπορικό σύστημα άντεξε στην κρίση. Φάνηκε αυτό κατά τη διάρκεια της ε, τελευταίας χρονιάς και αναδύεται ακόμα πιο ενισχυμένο έπειτα από αυτή τη δοκιμή αντοχής που υπέστη, η οποία κρίση ήταν και η πιο σημαντική μετά την τελευταία κρίση του 1998 που είχε πλήξει τότε τις ε, ε, πολύ δυνατές και αναδυόμενες τότε ασιατικές οικονομίες. Και μάλιστα ε, σε σύγκριση με την πέσινή κρίση, η κρίση του 1998 θεωρήθηκε πολύ μικρή. Τώρα, από εκεί και πέρα παρά τις μεγάλες αναταράξεις, τις πολύ ισχυρέ αναταράξεις, καταφέραμε να συνεχίσουμε την πορεία μας καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Βεβαίως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος των διαπραγματεύσεων, ωστόσο στα τελευταία 8 χρόνια διαπραγματεύσεων έχουν σημειωθεί μεγάλες πρόοδοι. Αναφέρομαι στη συμφωνία για την μπανάνα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λατινοαμερικανικών παραγωγών χωρών. Μια συμφωνία η οποία πλέον έχει έρθει προς ε, εξέταση εδώ σε εσάς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να τονίσω το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή και η κύρωσή της, η επικύρωσή της αν θέλετε από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σηματοδοτήσει και τη λήξη μιας πολιετούς διαμάχης και ως εκ τούτου θα δώσει νέα πνοή στον γύρο της Ντόχα. Τον περασμένο Δεκέμβριο έλαβε χώρα και η 7η Υπουργική Διάσκεψη και ήταν αυτή μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε όλη η οικογένεια του ΠΟΕ να εξετάσει από κοινού το σύνολο των δραστηριοτήτων της, τις συμφωνίες παρακολούθησης, τη βοήθεια σε αντάλλαγμα με το εμπόριο, Aid for Trade, την αναπτυξιακή βοήθεια, ε, τα διάφορα εργαλεία και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, μεταξύ άλλων. Αντίθετα με ό,τι πιστεύει η ευρύτερη κοινή γνώμη, ο ΠΟΕ δεν ασχολείται μόνο με τις διαπραγματεύσεις ε, του γύρου της Ντόχα. Βεβαίως αφιερώνουμε ε, χρόνο, δίνουμε πολιτική και τεχνική σημασία και προτεραιότητα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, έχουμε όμως και άλλες εξίσου σημαντικές δραστηριότητες. Τα μέλη του ΠΟΕ λοιπόν έλαβαν αυτό το σήμα, αυτό το μήνυμα, ότι δηλαδή ο ΠΟΕ λειτουργεί και μπορεί να λειτουργήσει. Άλλο σημαντικό τμήμα, άλλο σημαντικό σημείο τομής αν θέλετε ήταν η διάσκεψη της Κοπεχάγης για τις κλιματικές αλλαγές τον περασμένο Δεκέμβριο. Μια διάσκεψη η οποία κατέδειξε το ακαθόδες του θέματος αυτού. Εγώ δεν νομίζω ότι τα πράγματα πήγαν τόσο άσχημα όσο τα περιέγραψαν κάποιοι σε αυτή τη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Έχω τώρα μια κάποια εμπειρία, γνωρίζω πώς λειτουργεί η παγκόσμια διακυβέρνηση και για να είμαι ειλικρινής η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει άμεση σχέση με την, το περπάτημα του κάβουρα αν θέλετε ε, με πολλά βήματα εμπρός αλλά και οπισθοχωρήσεις συνάμα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει κανείς να επικρίνει τη διάσκεψη της Κοπενχάγης, ούτε να ε, περιορίζεται μόνο σε αυτήν καθεαυτή. Θα πρέπει να εξετάζει και τι έχει συμβεί έκτοτε με το πέρας ε, της ε, λήξη, με το της διάσκεψης της Κοπενχάγης. Αν δείτε σήμερα την κατάσταση θα καταλάβετε ότι περίπου 100 χώρες έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινοποίηση ή γνωστοποίησης. Δηλαδή συμπεριλαμβάνεται ε, σε αυτή την υποχρέωση το 80% των εκπομπών και αυτό είναι πρόοδος. Μπορεί να μην είναι αρκετή πρόοδος, είναι όμως πρόοδος. Θα ήθελα να ανατρέξω το παρελθόν και να μιλήσω για το, περίφημη ρίση του Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος είχε πει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί άπαξ μία φορά, αντιθέτως ε, θα οικοδομείται σιγά σιγά καθημερινά στο βαθμό που υπάρχουν συνέργειες και συμφωνίες μεταξύ των μελών ε, προκειμένου να υπάρξει κοινή πορεία προς τα εμπρός. Νομίζω ότι αυτό ισχύει περισσότερο παρά ποτέ σήμερα. Τώρα, το υπαριθμό ένα σημαντικό είναι η, ανάπτυξη, η ανάκαμψη. Και η ανάκαμψη είναι εφικτή μόνο όταν ε, αυξάνεται η απασχόληση. Μία ανάκαμψη χωρίς ε, αύξηση της απασχόλησης πυροδοτεί τα μέτρα προστατευτισμού αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλο και όλοι και αναγνωρίστηκε άλλωστε αυτό από το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο στην ε, Σύνοδο του Ντάλλας. Αυτά λοιπόν ε, συνιστούν τη μακροοικονομική εικόνα σήμερα ε, παγκοσμίω, εξού και παραμένει, ελοχεύει ο κίνδυνος του προστατευτισμού. Τι σημαίνει αυτό για εμάς στον ΠΟΕ ε, και για τις δραστηριότητές μας, τις οποίες εξετάζετε εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαίνει καταρχάς ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο τέλος του γύρου των διαπραγματεύσεων. Στο βόρειο τμήμα του πλανήτη εν υπάρχουν τα πιο σημαντικά πακέτα. Εκεί βεβαίως συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Σήμερα οι οικονομίες χρειάζονται όλο και πιο διαφορετικές πηγές οικονομικής μεγέθησης πέρα από, τα, ε, ε, πέρα από τις ενισχύσεις που προσφέρουν οι κυβερνήσεις. Επομένως, η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μπορούν η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να ε, στηρίξει την οικονομική μεγέθυνση και να συμβάλλει στην αύξηση και της απασχόλησης. Άλλωστε, διαπιστώνουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία από τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι δεν ολοκληρώνεται ο γύρος των διαπραγματεύσεων. Πολλές από αυτές τις χώρες δεν ε, ε, έχουν τα μέσα να ε, δώσουν τέτοιου είδους κίνητρα, κίνητρα τα οποία δίνουν ήδη οι ανεπτυγμένες χώρες. Είναι πολύ γνωστό ότι η υπομονή των αναπτυσσόμενων χωρών ε, εξαντλείται σιγά σιγά. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Συμφωνούν όλα τα μέλη και γι' αυτό το θέμα αυτό βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων μας. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε και τα ε, χρηματοπιστωτικά θέματα που έχουν να κάνουν με ε, το εμπόριο. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Παρακολουθούμε τον προστατευτισμό ως προς τις εμπορικές συναλλαγές. Από την άλλη όμως ε, παρακολουθούμε και το Aid for Trade διότι θέλουμε οι εμπορικές συναλλαγές, το εμπόριο, γενικότερα, να συμβάλλει στην ανάκαμψη. Θα πρέπει να υπάρξει συνθηκολόγηση μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας και των περιφερειακών ε, τραπεζών, αναπτυξιακών τραπεζών, ώστε να δημιουργηθούν διαβλή και κανάλια ε, επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε πολλούς τομείς τα επόμενα χρόνια και σίγουρα θα κληθούμε να τους συζητήσουμε ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, καλύτερη διάρθρωση μεταξύ του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Το η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη εμπειρία στο να εξισορροπεί αυτές τις δύο δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί πολύ καλά τη σύνδεση μεταξύ των εμπορικών συναλλαγών και των κλιματικών αλλαγών από την άλλη. Είναι θέματα που αρχίζουν και μας απασχολούν. Σε συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του ΠΟΕ και έχουμε ε, δημοσιεύσει ένα σχετικό έγγραφο για τα θέματα τα οποία θα έρθουν στο επίκεντρο της προσοχής μας στους επόμενους μήνες. Αυτά τα θέματα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας. Επίσης ε, η προσχώρηση νέων μελών του, ε, στον ΠΟΕ Έχουμε ξεκινήσει ορισμένες ε, διαπραγματεύσεις για προσχώρηση με ε, πολύ δύσκολη δουλειά η οποία γίνεται και από τους υποψηφίους και για τα ήδη ε, υπάρχοντα μέλη και πολλές από τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο ΠΟΕ έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις προσχωρήσεως. Ιδιαιτέρως αν σκεφτεί κανείς τι έγινε πριν μερικά χρόνια με την Κίνα για να προσχωρήσει. Πέραν αυτών υπάρχουν νέες θεσμικές ρυθμίσεις κατά τρόπον ώστε να αποφασίσετε και να αποδείξετε όχι μόνο ότι η Ευρώπη μιλά με μία φωνή, οπότε είναι και πολύ πιο αποτελεσματική, αλλά για να μπορέσει η Ευρώπη να συνεχίσει να ηγείται σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για αυτήν την ομιλία η οποία αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα από τις προσχωρήσεις νέων μελών στην ε, γενική θεώρηση του ΠΟΕ. Υπάρχουν πολλά σχόλια και ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. για τον κύριο Παπαστάμκο από το ΕΛΚ. Έχω, θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά έχω μια σειρά ερωτημάτων. Ε, πρώτο ερώτημα, αναφερθήκατε κύριε Γενικά, Γενικέ Διευθυντά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε τακτικός συνομιλητής ε, μαζί μας. Αυτό μας τιμά και χαιρόμαστε κάθε φορά που συναντώμεθα είτε εδώ είτε στη Γενέβη. Αναφερθήκατε στην πρωτοβουλία του G20 της Δευτέρας Απριλίου του 2009 στο Λονδίνο για την πολυμερή χρηματοδότηση του εμπορίου. Ήταν μια πρωτοβουλία. Ποια ήταν τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας γιατί προβλεπόταν και συγκεκριμένο ποσό για την ενίσχυση του, των εμπορικών συναλλαγών. Ε, δεύτερο επιμέρους ερώτημα ε, κυκλοφορούν φήμες ότι προσπαθείτε να αναδείξετε μια νέα προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις του γύρου της Δόχα. Αν θέλετε να παρακάμψετε, ε, να κάνετε bypass στις διαπραγματεύσεις, bypass από τα modalities για να, πάτε, για να πάμε στις ειδικέ δεσμεύσεις, τα scheduling specific commitments. Αν αυτό έχει κάποια βάση, ε, αναφερθήκατε επίσης στην παγκόσμια διακυβέρνηση και στη διάσκεψη της Κοπεχάγης για την κλιματική αλλαγή. Ανεξαρτήτως πώς αξιολογεί κανείς το αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης, μήπως θα επιβαρυνθεί η ε, η παγκόσμια εμπορική ατζέντα με περιβαλλοντικά θέματα ακόμη περισσότερο, ενώ εξορισμού άλλη είναι η αποστολή του, ε, του, WTO. Και ε, δυο τελευταία μικρά ερωτήματα σχετικά με τα αγροτικά. Ε, εκτιμάτε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα από τις αναδυόμενες οικονομίες να αναλάβουν δεσμεύσεις από τα emerging economies να αναλάβουν δεσμεύσεις στον τομέα των άμα και των υπηρεσιών. Και τέλος, πώς βλέπετε τον νέο ρόλο των ε, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ε, σε αυτόν τον γύρο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you from David Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο David Μάρτιν. Ε, κύριε Πρόεδρε, με τα χαρά σε βλέπω εδώ τον κύριο Λαμί, ιδίω όποτε έρχεται να συζητήσει μαζί μας. Τρία ερωτήματα έχω. Καταρχήν, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές διμερείς ε, διαπραγματεύσεις με, την, ε, με τον Καναδά, με την Κεντρική Αμερική, με διάφορες χώρες. Ε, πιστεύει ότι αν μπορεί να επιτύχει να συνάψει αυτές τις ε, εμπορικές συμφωνίες η Ευρώπη θα ε, προωθήσει την διεθνή οικονομία διότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από την Ιαπωνία να συνάψει μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κολλήσει όσον αφορά τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες και ίσως οι χώρες οι οποίες ε, δεν ε, συμμετέχουν σε διμερείς συμφωνίες θα ενδιαφερθούν περισσότερο για πολυμερείς. Ε, εσείς δηλαδή προς τα πού βλέπετε ότι πρέπει να κατευθυνθούμε. Επίσης συμφωνώ με ό,τι είπατε σχετικά με το εμπόριο και ίσως ε, δεν πρέπει να καταγγείλετε αυτούς οι οποίοι ε, δεν αποδίδουν αλλά ε, πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει κανείς ορισμένες χώρες να ευθυγραμμιστούν. Και τέλος, πιστεύετε ότι αν έχουμε ένα καλύτερο ορισμό της υποανάπτυξη χώρας θα μπορέσει αυτό να βοηθήσει στους στόχους μας, στην επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά διαγράψατε ένα πολύ ενδιαφέρον πανόραμα της διεθνούς κατάστασης αφενός όσον αφορά την κατάσταση κρίσης διότι υπάρχει μια διατροφική κρίση ήδη που προηγείται της οικονομικής ε, κρίσεως ε, και ε, που έπληξε περισσότερο τις χώρες που έχουν απελευθερώσει το γεωργικό τομέα αναφερθήκατε στην κλιματολογική αλλαγή, στην οικονομική οικονομική ε, κρίση ε, στις ε, διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τέλος αυτό που θα ήθελα να μου πείτε είναι ποιο είναι το συμπέρασμά σας από τις κρίσεις αυτές για τον ΠΟΕ και για τις απαιτούμενες προσαρμογές του. Διότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι ο ΠΟΕ έχει απομονωθεί στη διαπραγμάτευσή του και δύσκολα ε, ε, βγαίνει από αυτήν την, ε, την απομόνωση. Το πρώτο θέμα βέβαια το οποίο αναφέρθηκε ήταν ότι το εμπόριο και η απελευθέρωσή του θα ε, βοηθήσει ε, την ε, οικονομική απελευθέρωση αλλά βλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο ευάλωτες ορισμένες οικονομίες στους εξωτερικούς κραδασμούς και δι οικονομικούς. Επίσης Επίσης Εδώ μιλάμε για ε, μια φορολογία προσαρμογής στα σύνορα. Μια συζήτηση η οποία έχει γίνει. Ο επόμενος επίτροπος μετά από εσά ήδη σταμάτησε ε, αυτές τις σκέψεις, οπότε εσείς τι πιστεύετε. Αναφερθήκατε στην απασχόληση, στο κλίμα, αλλά όταν εξετάζουμε την πραγματική εργασία του ΠΟΕ και της διαδικασίες διαδικασίας διαπραγματεύσεως ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ του κύκλου της Ντόχα και των δικών σας στόχων. Ερώτησή μου λοιπόν, πόσο ο ΠΟΕ ε, θα ε, εντάξει αυτή την συστηματική κρίση, την διατροφική, την κοινοτική, την οικονομική, το πρόγραμμα διαπραγματεύσεως και στη διαδικασία διαπραγματεύσεως που παραμένει ένα σημείο άθικτο του ΠΟΕ όπου δεν, ε, δεν επηρεάζεται ούτε η μέθοδος εργασίας ούτε η, ο τρόπος διαπραγματεύσεως του ΠΟΕ για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ε, ε, συζητήσεις θα δώσω το λόγο τώρα εις τον κύριο Λαμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις ερωτήσεις του κύριου Παπαστάμκου, πρώτα απ' όλα. Για το τμήμα της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, Trade Finance, όπως είπα και πριν, παρά την κρίση, είχαμε και μείωση της ζήτησης του διεθνούς εμπορίου αλλά και το σοκ το οικονομικό συγχρόνως που ορισμένοι αποσύρθηκαν πλήρως από την αγορά. Πράγμα το οποίο δημιούργησε, συνεισέφερε στην κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου. Σε τι βαθμό η εκτίμηση λέει 10 με 20% της μείωσης της περσινής προκλήθηκε από ένα καθαρά δημοσιονομικό πρόβλημα. Και σε αυτό αντιδράσαμε, όχι μόνοι μας εξάλλου, όχι μόνο εμείς. Δημιουργήθηκε ένα λόμπι, ήμασταν εμείς επικεφαλής, με τους φίλους μας από τράπεζες και την Περιφερειακή Τράπεζα Ανάπτυξη, την Αφρικανική, την ε, Αμερικανική, την Ένωση της Βέρνης, όπως συμμετέχουν εξαγωγείς και φτιάξαμε αυτό το πακέτο των 150 δις δολαρίων που εγκρίθηκε στο Λονδίνο που ήταν ένα πακέτο ρευστού χρήματος. Από τότε φτιάξανε κάπως τα πράγματα. Η προσπάθεια, η δημόσια έφερε αποτελέσματα. Συγχρόνως είδαμε και στη δικιά μας την πτυχή βελτιώσεις όσον αφορά το θέμα του κινδύνου εντάξει η ρευστότητα, αλλά μετά υπάρχει ακόμα κίνδυνος αρκετά υψηλός και ακόμα και αν μειώθηκε από πέρυσι, παραμένει σε επιλεκτικό επίπεδο. Μικρές χώρες ή χώρες λιγότερο αναπτυγμένες, οι μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται πολύ. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες λοιπόν με όλους τους εμπλεκόμενους πριν από τον Ιούνιο τους G20 κάπου στον Απρίλιο δηλαδή, και από την άλλη έχουμε και συζητήσεις που δεν είναι όλες δημόσιες και ανοιχτές, έτσι, με τις ρυθμιστικές ε, δημοσιονομικές αρχές σε διεθνές επίπεδο, οργάνωση στην Βασιλεία με την Επιτροπή της Βασιλείας αλλά και της Δημοσιονομικής Σταθερότητας έχουμε συζητήσεις, αρκετά περίπλοκες βέβαια. Πολλοί, όπως και εγώ, πιστεύουμε ότι οι ρυθμιστές έχουν την τάση να μπερδεύουν ε, τα πράγματα, δηλαδή ε, να βάζουν να μπερδεύουν με τα τοξικά δάνεια τα οικονομικά και να υπάρχουν και κεφάλαια κινδύνου. Εγώ δεν λέω ότι μπορώ να κάνω θαύματα, έτσι κι αλλιώς έχουμε συγκεκριμένη εντολή. Πάντως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία, δηλαδή είναι όπως όταν χτίζεται ένα κτίριο ξεκινάμε από ένα αρχιτεκτόνημα και σιγά σιγά βλέπουμε ποιες είναι οι δυσκολίες, περνάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μετά καλούμε μια επιχείρηση, ε, μετά καλούμε τους ε, εργολάβους, τους ε, εργάτες, σιγά σιγά βλέπουμε πώς προχωράει και τελικά βάζουμε και τετραυλικά, τα ηλεκτρικά και βάφουμε και το κτίριο στο τέλος. Έτσι προχωράμε, σιγά σιγά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κάνουμε βραχικύκλωμα, πρέπει να περνάμε από όλα αυτά τα στάδια. Και όντω είμαστε σε ένα στάδιο που έχουμε το κτίριο, υπάρχουν κάποια κυκλώματα εσωτερικά τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε πόση ενέργεια ακριβώς θα χρειαστεί το κτίριο για να λειτουργήσει. Μας λείπει δηλαδή το δεδομένο της πολιτικής ενέργειας, άμα θέλετε. Εντάξει, τα καλώδια, εντάξει, οι μπρίζες, αλλά χρειάζεται όλα αυτά να τα βάλουμε να δουλέψουν. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το στάδιο. Περιμένουμε να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πολιτικό περιεχόμενο της συμφωνίας. Για να μην έχουμε μετά να ετοιμάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, είμαστε στο τέλος στο τελείωμα. Δεν πρόκειται για βραχή κύκλωμα, πρόκειται για σχεδιασμό του τελειώματος του κτηρίου που πρέπει να γίνει έγκαιρα. Για την γεωργία τώρα. Είναι αλήθεια ότι οι αναδυόμενες χώρες, αναδυόμενες οικονομίες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στις γεωργικές διαπραγματεύσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Έχουμε ακόμα τη ρήτρα διασφάλισης για τις υπονάπτυξη χώρες σε περίπτωση μεγάλων εισαγωγών. Σίγουρα οι χώρες αυτές έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και όχι μόνο η Βραζιλία και είμαστε σε μια κατάσταση σήμερα που είναι πιο ξεκάθαρη μετά την κρίση παρά πριν από την κρίση. Είμαστε λοιπόν λέω σε μια κατάσταση όπου οι δεσμεύσεις από τις διάφορες υποανάπτυξη λοιπόν, χώρες όσον αφορά την τελική συμφωνία ποικίλουν περισσότερο από ό,τι πριν, νωρίτερα. Ξέρετε ότι τώρα στην οικονομική σκηνή και εμπορική διεθνή ε, σκηνή έχουμε τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα, την Ινδονησία, την Νότια Αφρική, την Αίγυπτο. Οι γίγαντες, κατά κάποιο τρόπο, των οποίων η συμβολή όσον αφορά την λειτουργία της διεθνούς οικονομίας είναι χωρίς σύγκριση με το, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δεν μπορεί να ζητάτε τα ίδια από την Κίνα, την Ινδία, όπως ζητάτε από την Βουργίνα Φάσο, την Κένια, την Καμπότζη. Υπάρχει διαφοροποίηση στην ε, συνεισφορά. Γίνεται, προγραμματίζεται ήδη και μερικές φορές πολιτικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν συνήθειες. Το παιχνίδι ήταν φοράς βορράς-νότος. Ε, τώρα πια δεν είναι έτσι. Τώρα έχουν αλλάξει οι συνθέσεις των ομάδων. Έπειτα οι ίδιες οι αναδυόμενες οικονομίες το αναγνωρίζουν. Για να ε, δούμε το θέμα της ε, βοήθεια στο εμπόριο. Εκείνοι που πρέπει να βοηθάνε τις λιγότερο προηγμένες χώρες, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική πρόοδο, είναι σήμερα και η Κίνα και η Ινδία και η Βραζιλία με μια ιδιαίτερα δραστήρια πολιτική στην Αφρική. Η Κορέα μπαίνει σε αυτό το δρόμο. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση σήμερα η οποία αναμφίβολα θα επηρεάσει το όλο σκηνικό. Προς τον David Μάρτιν τώρα. Ναι, μίλησες για stumbling blocks, δηλαδή τις δυσκολίες, τις μεγάλες. Ναι, είναι μια συζήτηση αυτή η οποία έχει απασχολήσει ακαδημαϊκούς για δεκαετίες και δεκαετίες. Και έχουν γραφτεί όγκοι άρθρων, τόμοι άρθρων είναι ένα ζήτημα που βάζει πολλούς να σκεφτούν. Πάντως η άμεση απάντηση στην ερώτησή σου είναι εξαρτάται. Εξαρτάται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι διμερείς ε, συζητήσεις μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου Ισχύει το αντίθετο. Θα ήταν κακό. Η περιφερειακή ολοκλήρωση, για παράδειγμα, που παίρνει την μορφή δημερών συμφωνιών, έχει αποδειχτεί κάτι θετικό. Το κάναμε παλιά. Και καλό στις χώρες ΑΣΕΑΝ σήμερα. Είναι θετικό τι γίνεται σε υποπεριφέρειες στην Αφρική. Και εκεί είναι θετικό, στην Αμερική. Τώρα όμω, οι προϋποθέσεις είναι βασικά ότι αυτές οι διμερείς συμφωνίες είναι ένα θετικό για τον ΠΟΕ. Προσθέτουν κάτι παραπάνω. Πράγματι, υπάρχουν κάποιες αρνητικές συνέπειες Ιδίω επειδή είναι περίπλοκες οι διαδικασίες, γιατί όταν δώσετε την προτίμηση σε μια χώρα πρέπει να ε, αποδείξετε την προέλευση κτλ. Όλα αυτά κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Έτσι λοιπόν, de facto, και αυτό είναι που κοιτάμε πολύ προσακτικά και αναλύουμε αυτή την εποχή, η πραγματικότητα είναι ότι η αναλογία αυτών των διμερών ε, προτιμήσεων που υπάρχουν και που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις είναι τελικά μικρή. Τάξη μεγέθους από τα στοιχεία που έχουμε είναι 30-40%. Οπότε η απάντησή μου στην ερώτηση είναι ότι πρέπει να δούμε σε τι βαθμό ισχύει στην πραγματικότητα πριν πάμε πίσω στο πρόβλημα της αρχικής αρχιτεκτονικής. Τώρα, προς το παρόν, έχουμε στοιχεία τότε που ο Gordon Brown πίεζε πολύ. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά έχουν τηρηθεί. Μπορεί να είναι μια περίεργη ιστορία αυτή, γιατί οι διεθνέ εξελίξει ε, όσον αφορά την αλλαγή. ήταν. Αλλά αυτή η βοήθεια για το εμπόριο προς το παρόν, Aid for Trade, λέει ότι οι υποχρεώσει έχουν συμπεριληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα θυμόσαστε ότι ήταν 50% από τα κράτη-μέλη και 50% από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Τα στοιχεία αυτά τα αναθεωρήσαμε πέρυσι με την αναθεώρηση που κάναμε στο Aid for Trade, με διάφορους διεθνείς οργανισμούς που προσπαθήσαμε να συντονίσουμε και τότε ήταν εντάξει τα στοιχεία. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μια νέα global review, μια νέα αναθεώρηση, όπου να είναι, και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Φέτος δεδομένων των δημοσιονομικών ε, περιορισμών και μετά από τα καλά αποτελέσματα, τι θα δούμε. Θα δούμε ότι επιβεβαιώνονται και φέτος αυτά τα καλά αποτελέσματα. Η θα σας πείσω περισσότερα γιατί εκείνη τα έχει αυτά τα θέματα. Αν πάντως εντοπίσουμε εκεί ότι κάτι δεν πάει καλά, να ξέρετε ότι πολύ γρήγορα θα ξανάρθουμε. Εκείνη, εγώ γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή όπου, όπως είπα, αναπτυσσόμενες χώρες διαπιστώσουμε ότι γίνονται θύματα, αν τα δημοσιονομικά δεν πηγαίνουν καλά, σίγουρα δεν πρέπει δύο φορές να τιμωρούνται για την κατάσταση αυτές οι χώρες. Και για την τελευταία ερώτηση, David. Κοίτα, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέο ορισμό για το τι είναι μία αναπτυσσόμενη χώρα. Εκτός αν χρειαζόμαστε και ένα νέο ορισμό για το τι είναι θεμητό εμπόριο, δίκαιο. Η πραγματικότητα, η ομή πραγματικότητα είναι ότι το σύστημα των διεθνών εμπορικών ρυθμίσεων, το σημερινό, υπάρχει από τη δεκαετία του 90, τότε που η ισορροπία δυνάμεων ήταν διαφορετική. Και χρειάστηκαν χρόνια ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να φτάσουν στο σημείο να πούνα γιατί φαντουργία και ρουχισμός» Εκεί είχαν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις πλούσιες χώρες. Με την ίδια λογική χρειάζονται και χρόνια για να γίνεται το ίδιο στη Γεωργία. Ο γύρος της Δόχα δεν είναι παρά μία κίνηση προκειμένου να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο υποχρεώσεων και πλεονεκτημάτων και μερικές φορές η κίνηση αυτή είναι περίπλοκη, είναι δύσκολη. Οπότε αν ολοκληρωθεί ο γύρος, 80% των αποτελεσμάτων τα έχουμε. Αν λοιπόν ολοκληρωθεί, θα είναι υπέρ της ανάπτυξης, διότι θα ενισχύσει την πειθαρχία σε τομείς όπως είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις, οι εξαγωγών, που έκαναν κακό στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους και θα δημιουργήσει ένα σύστημα που θα είναι πιο δίκαιο. Αυτό είναι το στοιχείο το αναπτυξιακό στον γύρο αυτό της Δόχα. Γενικ Ζαντό τώρα. Με ρώτησε πολλά πράγματα. Κοίταξε, η κρίση υπάρχει και ο ΠΟΕ κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα λε. Με την ίδια μερίσια διάταξη, τη γνωστή. Γιάννικ, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από την αρχή της κρίσης, πρέπει να πω και έχω εδώ και άλλους που μπορούν να το πούν επίσης και άλλα μέλη του ΠΟΕ, ότι από την αρχή της κρίσης αυτής έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αν μην τι άλλο κινητοποιήθηκαμε φοβερά σε αυτό το θέμα του ελέγχου. Και το σύστημα ΠΟΕ δεν έμεινε αδρανές, όχι, αντίθετα. Δραστηριοποιηθήκαμε και μάλιστα ακριβώς επειδή κινητοποιηθήκαμε, και βάσει της πειθαρχία που υπάρχει καταφέραμε να αντισταθούμε σε αυτό το προστατευτισμό. Αν δείτε στα τέλη του 2008 τι γράφανε εφημερίδες, ξεκινάμε με ένα νέο κύμα προστατευτισμού. Ε, λοιπόν όχι. Και δεν λέω ότι είναι μόνο το σύστημα του ΠΟΕ και εμείς που φροντίσαμε, υπήρξε και μια αλλαγή στην οτροπία γενικότερα, η οποία μας οδήγησε εκεί που είμαστε σήμερα. Γιατί πια ξέρουμε ότι αν αρχίσουμε προστατευτισμό, εμείς, ε, οι άλλοι τι θα κάνουν, το ίδιο. Και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο. Τώρα υπάρχει αλληλοεξάρτηση. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα πού βρισκόμαστε. Έχουμε νέες εξελίξεις. Περιβάλλον. Είμαστε στη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Έχουμε μια συγκεκριμένη εντολή. Από τα 20 θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη του γύρου υπάρχει ένα που είναι σε θέματα ανοίγματο ανταλλαγών δίνουμε πλεονέκτημα όταν πρόκειται για αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον. Περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες. Θα είναι στα συμπεράσματα. Καταλαβαίνει κανείς, δεν είναι δύσκολο, ότι τι είναι περιβαλλοντικό αγαθό και περιβαλλοντική υπηρεσία, αυτό μπορεί να επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνισμού που έχει ο καθένας και τι θέλει από τους ε, ανταγωνιστές και τέρους του. Είναι λογικό. Αν ε, λέει κάποιος ότι έχει ξαναπλυντήριο, ότι από χρησιμοποιεί νερό, τι είναι, ε, η εντολή πάντως αυτή είναι και προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Για θέματα τώρα τροφίμων και ασφάλειας διατροφικής. Συμμετέχουμε, συμμετέχω και εγώ στην ε, Task Force και ένα άλλο αναπληρωτή μου επίσης, επιμονή μου βάσεω ασχολείται με αυτό το θέμα και συμμετέχουμε. Είναι μια δύσκολη συζήτηση. προσπαθούμε να δούμε πιο ξεκάθαρα. Οι διεθνείς συναλλαγές και η διατροφική κρίση σε τι σχέση βρίσκονται. Και ο ΦΑΟ, και το στη Ρώμη, η ανάπτυξη του ΟΗΕ κλπ. Όλοι μαζί λέμε ότι χρειάζονται συναλλαγές ανοιχτές στο γεωργικό τομέα ώστε να διευθετηθεί το θέμα αυτό της διατροφικής ασφάλειας. Έχουμε κάποιες καλές ιδέες. Ένας από τους λόγους για τους οποίους βρεθήκαμε σε αυτή την κρίση, και δεν είναι βέβαια και ο μόνος, είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν φοβερά και ανεβαίνουν για λόγους και δημογραφικούς και γεωγραφικούς, αλλά και για λόγους ανάπτυξης γιατί το μείγμα αυτού που κερδίζει 50-20 δολάρια είναι διαφορετικό. Δηλαδή τι τρώει αυτός από αυτόν που παίρνει ένα δολάριο την ημέρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και γι' αυτό πρέπει να βελτιωθεί η σχέση προσφοράς και ζήτησης. Το διεθνές εμπόριο είναι εμπόριο. Είναι ο καλύτερος τρόπος συναλλαγής με τον τρίτο κόσμο. Εκεί που υπάρχουν ε, πολλά εξάγουμε και εκεί που υπάρχουν λίγα εισάγουμε. Και όταν υπήρξε απόφαση για να σταματήσει η παραγωγή δημητριακών, ε, κάπου ήταν γιατί υπήρχε τεράστιο πλεόνασμα ενώ είχαν λίγο νερό. Οπότε απευθυνθήκα στο διεθνές εμπόριο για να μπορέσουν να εισάγουν ό,τι δεν μπορούσαν πια να παράγουν οι κανόνες του παιχνιδιού στο διεθνές εμπόριο για τη Γεωργία πρέπει να είναι πιο σωστοί. Έτσι απαντάω στην τελευταία ερώτηση του David πριν. Έρχομαι τώρα στον φόρο, στα σύνορα. Φυσικά και ο ΠΟΕ ξέρει ότι γίνεται αυτή η συζήτηση δεξιά και αριστερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, αν και μόλις ξεκίνησε. Το Αμερικανικό Κογκρέσο γίνεται. Έχει ξεκινήσει μόλις. Κοιτάξτε για μένα, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Γενικά μιλώντας, ένα τέτοιο φόρος, ένα τέτοιο τέλος, είναι καλό ή όχι. Αν εγώ έδινα απάντηση σε αυτό, θα μου παίρνω το κεφάλι οι νομικοί, αλλά και οι περισσότεροι από τον ΠΟΕ. Οπότε γι' αυτό η απάντησή μου είναι εξαρτάται. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλους, καταρχήν να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, βάλαμε επιτάπητος μία έκθεση από κοινού ΟΗΕ και ΠΟΕ, προκειμένου να δούμε αυτό το παζλ. Έχει όλα του τα κομμάτια. Το αποτέλεσμα προς το παρόν είναι ότι δεν υπάρχει κόκκινο φως, αλλά ούτε και πράσινο φως. Ούτε ναι, ούτε όχι. Πρέπει να δούμε κατά περίπτωση. Πρέπει να αναρωτηθούμε, για παράδειγμα, τι θα εξυπηρετούσε ένας τέτοιος φόρος ε, καυσίμων στα σύνορα. Αν πρόκειται για τον άνθρακα. Πρέπει να δούμε. Ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ και από τους πιο σπουδαίους περιβαλλοντολόγους ή κλιματολόγους. Και πώς μπορεί κανείς να υπολογίσει το ίχνος άνθρακα μιας εισαγωγής. είναι σε μερικές περιπτώσεις το ίχνος αυτό καλύτερο από εκείνο της ε, παραγωγής εντός των συνόρων. Και τι κάνετε μετά. Πώς γίνεται ο υπολογισμός ακριβώς. Είναι περίπλοκο και πρέπει να καταλάβουμε όλη τη λογική που βρίσκεται από πίσω. Πάντως η απάντηση δεν είναι τόσο τεχνική, η απάντηση είναι πολιτικής φύσεως. Δηλαδή θα έχουμε ένα σύστημα πολυμερές τύπου Κοπεχάγης, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι για λόγους τόσο ιστορικούς όσο και πολιτικούς, η φύση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, οι Άπωνες από τη μία και από την άλλη μεριά ε, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία κλπ. δεν μπορεί να είναι ίδια. Είναι πολιτικοί λόγοι. Ή λοιπόν που θα έχουμε κάτι όπου όλοι θα συμφωνήσουν ότι θα πάρουμε αυτή την κατεύθυνση, αλλά με διαφορετικά μέσα ο καθένας και τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε θέματα εμπορίου ή δεν θα το κάνουμε αυτό και τότε κινδυνεύουμε να έχουμε προβλήματα. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι έτσι γιατί μου ήρθε. Είναι θέμα εμπειρίας. Αν δούμε τι έχουμε από συμφωνίες πολυμερείς μέχρι σήμερα Πολλές από τις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν εμπορικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς συμβάσεις για τα τοξικά, για προστατευόμενα είδη, το πρωτόκολλο του Μόντρελ, για τα, τον χλωροφθοροάθρακα. Είναι η Διεθνή Συμφωνία που έχει υπογραφεί από τους περισσότερους ποτέ. 196 υπογραφές, ρεκόρ. Η συμφωνία αυτή περιλάμβανε εμπορικά μέτρα και περιλάμβανε και μέτρα διορθωτικά, αλλά όχι εμπορικές κυρώσεις. Άρα μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι πολιτική. Αν χρειάζονται εμπορικές διορθώσεις μέσα εμπορικής πολιτικής, αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη για μια πολυμερή συμφωνία. Αυτή χρειάζεται. Αν έχουμε μια σωστή συμφωνία, προβλέπω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί όσοι έχουν συνυπογράψει και αναγνωρίζουν την ανάγκη σε ένα τομέα, θα κάνουν το ίδιο και σε ένα άλλο τομέα που είναι εμπορικέ συμφωνίε. Ευχαριστώ. Έχω πολλούς που ζητούν το λόγο και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα έχουμε 25 λεπτά ακόμη. Οπότε για να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο των πολιτικών ομάδων ξεκινώντας με τον εκπρόσωπο των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ως και εισηγητής για το ψήφισμα στο Κοινοβούλιο θα ήθελα καταρχήν εν ονόματι των φιλελευθέρων να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ αλλά επίσης και ε, για το ότι στην 7η Υπουργική Διάσκεψη σταθήκατε ε, στο πλευρό μας και η συνεργάτη σας ε, έτυχε όλη της ευγνωμοσύνης μας. Αναφερθήκατε σε ένα θέμα, ότι ο ΠΟΕ απέδειξε τις δυνατότητες του ή στην κρίση. Εάν δεν υπήρχε ο ΠΟΕ θα έπρεπε να το έχουμε εφευρέσει τώρα και γι' αυτό μπορέσαμε να αποφύγουμε ε, μία κλιμάκωση ε, προστατευτισμού. Και εδώ αναφερόμαστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παντού διεθνώς και βλέπουμε ότι τα πολυμερή συστήματα από τη γνώμη μας είναι πολύ πιο σημαντικά και αποδοτικά από ότι οι διμερείς συμφωνίες για να μπορέσει κανείς να προωθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από την πολιτική και οικονομική κρίση θα υπάρξει μία πιο ψύχρεμη θεώρηση του παγκοσμίου εμπορίου, το οποίο δεν ε, ευθύνεται ε, για όλα τα προβλήματα του κόσμου αλλά δεν είναι και πανάκια. Ε, χρειάζεται ένας, μια ρεαλιστική αισιοδοξία ή μια αισιόδοξη ρεαλιστική θεώρηση. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε για τις οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν στις συσκέψεις στη Γενέβη έχουν αντιληφθεί διαφορετικά τώρα της τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα. Έχετε απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν βασικό παίκτη στα θέματα των τωρινών διαπραγματεύσεων, διότι δεν μιλάμε μόνο για λίγους μήνες μετά από την ολοκλήρωσή τους, αλλά εμείς και όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου αποδεικνύοντας το από το ψήφισμά τους έχουν μεν συγκεκριμένες επιθυμίες αλλά και εσείς θα θέλατε κάτι από την Ευρώπη. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι χρειάζεται για να μπορέσει ε, να απεγκλωβιστεί το μεγάλο πλοίο της Ντόχα από το σημείο στο οποίο έχει παραμείνει. Ευχαριστώ. Τώρα ο ο Ρόμπερ Στέρντι. Θα είμαι πολύ σύντομος σε ότι των ε, Βρετανών συντηρητικών. Ε, όταν μιλήσαμε για διμερή και πολυμερή, πιστεύω όπως και ο Ντέιβιτ ότι οι, πολυ... διμερείς μπορεί να καταλήξουν σε πολυμερείς συμφωνίες όπως είπατε άλλωστε στα λεγόμενά σας. Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκεται τώρα η κατάσταση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τις χώρες Μερκοσούρ. Υπάρχουν διμερείς ε, συμφωνίες, ε, υπάρχει η προοπτική να προσχωρήσουν εις ε, το ΠΟΕ και να δεχθούν αυτά που λέτε. Ε, αλλά αν όχι, γιατί θεωρούν ότι δεν είστε αρκετά σημαντικός, ε, θα πρέπει να ε, φτάσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων των Αμερικανών την τελευταία στιγμή να δεχθούμε ό,τι μας επιβάλλουν για τις ταινίε, για όλα τα προϊόντα, τα πάντα και νομίζω ότι δεν έχουμε καλή διαπραγματευτική θέση αυτή τη στιγμή. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε, διαπραγματεύουμε, ε, διαπραγματευόμαστε τώρα με τις Ηνωμένε Πολιτείε ή περιμένουν τις εκλογές για το Κογκρέσο. Και τέλος, ο Χέλμουτ Σούλτς από το Ινγκούεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και κύριε Γενικέ Διευθυντά. Στην αρχή ε, ε, είχα ρωτήσει από διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, εν ώψη αυτής της συζητήσεως τι ερωτήσεις θα είχαν ε, από την ομιλία σας και μου είπαν ότι δεν περιμένουν τίποτα διότι πιστεύουν ότι δεν έχει κανείς να προσθέσει πολλά στον τωρινό ρόλο του ΠΟΕ. Θεωρώ όμως αυτή τη θεώρηση πολύ, πολύ απεσιόδοξη. Ε, είπατε ε, για το κτίριο το οποίο οικοδομείται με το γύρο της Ντόχα και ίσως θα έπρεπε ε, να διερευνήσουμε λίγο περαιτέρω. Δηλαδή το οικοδόμημα το οποίο οικοδομείται όπου δεν λειτουργούν όλα καλά αυτή τη στιγμή ε, μπορεί να αποτελέσει ένα μελλοντικό στοιχείο ή ε, η πρόσωψη θα είναι τόσο άσχημη ώστε κανείς δεν θα θέλει να μπει μέσα. Δηλαδή πώς εσείς αξιολογείτε δείτε την θέση των ΗΠΑ για να συμβάλλουν σε μία αναθεώρηση του διεθνούς εμπορικού συστήματος ή ε, ε, πρέπει να παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο ο ΠΟΕ. Επίσης, δεύτερη ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας, πόσο θα ήταν δυνατόν να υπάρξει μία πιο αυστηρή διεκπαιρέωση αυτών των ε, διαπραγματεύσεων κατά τρόπον ώστε να αποδείξουμε ε, ότι οι ε, προχωρημένες χώρες και ανεπτυγμένες χώρες καταστρέφουν με τις πράξεις τους την ε, πρόοδο του διεθνούς εμπορίου. Έχει λεχθεί ότι η εκθετική πρόοδος θα μπορέσει να οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο. Είναι σωστό όμως αυτό. Ε, ρωτώ, Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον ΠΟΕ την μελλοντική πολιτική κατά τρόπον ώστε η κοινωνική πολιτική, η κλιματολογική πολιτική να μπορέσουν επίσης να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Κύριε Λαμή, ε, νομίζω ότι τώρα πρέπει να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και θα ήθελα να μας διαθέσετε λίγο χρόνο γιατί υπάρχουν ακόμη πολλοί που έχουν εγγραφεί για να σας κάνουν ερωτήσεις. Ωραία, κατάλαβα και το σημειώνω. Όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Τόιρερ, καταρχήν, ξέρω ότι υπήρξε πάντοτε μεγάλη ευαισθησία σε αυτή την ε, Επιτροπή ε, για το διεθνές εμπόριο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πολύ σωστά, διότι σε πολλούς τομείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ουσιαστικά ο ιστός του διεθνούς εμπορίου. όχι τα μεγάλα διεθνή ονόματα και εταιρείε, αλλά αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μία ειδική συμφωνία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των εμπορικών διευκολύσεων που εάν ολοκληρωθεί θα μπορέσει να οδηγήσει σε μία μεγάλη διευκόλυνση και απλούστευση των απαιτήσεων για να μπορεί κανείς να υποφεληθεί από το διεθνές εμπόριο. Έχουμε μία μελέτη του Ινστιτούτου Πίτερσον στην Αμερική που λέει ότι ε, τα ωφέλη του γύρου στους άλλους 19 τομείς θα διπλασιαστούν εάν μπορέσουμε να περιλάβουμε στις διαπραγματεύσεις το 20 αυτό στοιχείο που είναι οι εμπορικές διευκολύνσεις. Διότι για πολλές χώρες η ε, πρόσβαση στο διεθνές εμπόριο είναι πάρα πολύ δυσχερής λόγω των τελωνιακών διατυπώσεων και εμπορικών μεθόδων όσον αφορά το εμπόριο σε σχέση με πριν από 6-10 ε, χρόνια πριν. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει πιο σημαντική συζήτηση και πιο ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή, στο παρελθόν, στις συζητήσεις μας υπήρχαν ε, παρανοήσεις που τώρα έχουν εξαφανιστεί. Βέβαια, με ορισμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όχι όλες, και δεν θέλω εδώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα, διότι δεν νομίζω ότι είναι προς όφελός τους. Έχουμε μία σχέση σαν με τις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δηλαδή, ε, με ορισμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουμε συζήτηση ε, παραδείγματο χάρη θα μας στηρίξετε αν επιτύχουμε το τάδε ε, αποτέλεσμα δηλαδή είναι μια ενεργή πολιτική διεργασία ενώ με άλλες είναι πολύ διαφορετική κατάσταση Παραδείγματο χάρη όσον αφορά το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τώρα ε, γίνεται πιο ανοιχτή συζήτηση σε πιο δημόσιο χώρο. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά ε, το θέμα αυτό, τη συμπεριφορά μου, τη συμπεριφορά των βοηθών μου και της γραμματείας, επηρεάζεται από την ευαισθησία πολλών μελών μας. Αλλά προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσει να επιτύχει κανείς σε καλύτερη αλληλεπίδραση. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Δύο πράγματα. Καταρχήν θα πρέπει ο ΠΟΕ να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο δεν πρόκειται να είναι όπως πριν από 10-15 ε, χρόνια και βλέπω κάποιον να μηδιά στο βάθος της ε, ε θούσης, αλλά τότε η ε, ε, Ευρώπη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδά και η Ιαπωνία μαγειρεύανε κάποια λύση και μετά έστελναν επιδέξιους διπλωμάτες να το πουλήσουν στους υπόλοιπες χώρες του ο κόσμο. Αυτό δεν γίνεται ε, πλέον. Υπάρχει η Κίνα, η Βραζιλία, οι Αφρικανικές χώρες, οι χώρες ΑΚΕ και εδώ αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε ηγεσία. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηγεσία από ό,τι στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το δεξαμενόπλιο διότι αυτό είμαστε όχι ένα μικρό πλιαράκι της ακτοφυλακής ε, δεν είναι αυτό ο χαρακτηρισμός ο σωστός χρειάζεται το μεγάλο αυτό πλοίο να έχει έναν προβλέψιμο και ουσιαστικό ηγέτη στις διαπραγματεύσεις. Και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και την ουσία τους υπάρχει ένας τομέας όπου θα ήταν προς όφελος όλους από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να έχουμε μία πιο σαφή και δραστήρια πολιτική και αναφέρομαι εδώ εις τις επιδοτήσεις της αλίας. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, αλλά στη θέση σας, σε αυτή την Επιτροπή, και αντιλαμβάνομαι ότι η άποψή σας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επηρεάζει τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ε, πιστεύω ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας θα έπρεπε να πιέσουν τα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ρόμπερτ. Όσον αφορά την απλή απάντηση στην ερώτησή σου, πρέπει να σου πω ότι δεν ξέρω, διότι εγώ δεν συμμετέχω σε διμερείς ε, διαπραγματεύσεις, ούτε πρέπει να, να συμμετέχω. Οπότε, ε, πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μερκοσούρ, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Όσον αφορά τις ε, ε, Ηνωμένε Πολιτείε και το Μερκοσούρ εάν ε, διαβάζω σωστά τις εφημερίδες δεν ε, είναι πολύ δραστήριο το μέτωπο δραστήριο μέτωπο είχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Κολομβία αλλά υπάρχει ένα σχέδιο που ακόμη δεν έχει υποβληθεί στο Κογκρέσο προς επικύρωση. Το ερώτημα λοιπόν είναι... Οι Ηνωμένε Πολιτείε ενδιαφέρονται, εγώ θα σας πω ναι. Ξέρω ότι όλοι δεν συμφωνούν ε, με αυτή την άποψη ε, όσον αφορά τα μέλη του ΠΟΕ. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω διότι μόλις υπάρξει μια διαφορετική διάγνωση, εάν η Γενική Διεύθυνση λάβει διαφορετική θέση, ε, εμφανίζομαι σαν να αποκλίνω από την ουδετερότητά μου. Αλλά μιλώντας σε ειδικού σαν και σας, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι ιδίω όσον αφορά την τελευταία δήλωση του Προέδρου προς το Κογκρέσο αρχίσαμε να βλέπουμε ένα διάγραμμα του τι σκοπεύει να κάνει αυτή η διοίκηση της ε, ε κυβέρνησης Ομπάμα η οποία θέλει να βγει από την κρίση, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να αυξήσει τις εξαγωγές όχι μόνο με ε, διαφορά ρετικά επίπεδα ανάπτυξης, παρόλο που και αυτό θα είναι ε, απαραίτητο αν ε, σκεφτεί κανείς πώς θα εξελιχθούν οι εξαγωγές στο μέλλον. Αν δείτε την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τις διάφορες χώρες, ε, υπάρχει ε, μία, ένας διαφορετικό επίπεδο ρόλου και αυτό συμβάλλει στις εξαγωγές. Άρα οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εκτεθειμένες, εμπλέκονται και προσπαθούν να διαπραγματεύσουν και αυτό είναι κατανοητό διότι στο εσωτερικό είχαμε, ε, είχαμε αμφιβολίες για το τι προσφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και ε, μέχρι την τελευταία στιγμή θα σας λέμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι δεν, δεν, δεν βγαίνουν τα κουκιά, αλλά ουσιαστικά όσον αφορά την ουσιαστική στρατηγική δεν ξέρω τι γίνεται και αν ήξερα πάλι δεν θα μπορούσα να σας το πω. Εσείς πρέπει να το μαντέψετε μόνοι σας. Προς τον κύριο Σούλτς. Σόλτς. Η, ε, πολιτική αλήθεια αυτού του οικοδομήματος το οποίο ανέφερα προηγουμένως είναι ότι στην αρχή το 2001 υπήρχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρώπη που έσπροχναν και ο ΠΟΕ και οι υπόλοιπες χώρες που ακολουθούσαν χωρίς μεγάλο ενθουσιασμό. Δέκα χρόνια όμως αργότερα έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Ποιος πιέζει περισσότερο για να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα ε, είναι υποανάπτυκτης χώρες και αυτό για πολλούς λόγους καταρχήν ε, την κατάσταση της παγκοσμίου οικονομίας, ε, το τι πρόκειται να βοηθήσει την Ευρώπη και την ανάπτυξή της αλλά ουσιαστικά βλέπουμε ότι όσο αναπτυσσόταν η διαπραγμάτευση άλλαξαν οι παίκτες και ε, γι' αυτό θέλω να απαντήσω και στον κύριο Στέρντι ότι νομίζω ότι οι χώρες ενδιαφέρονται ότι θέλουν να υπάρχει ε, ένα σύστημα κανόνων πολυμερών και όπως όλες οι οικονομίες που είναι πιο ανοιχτές από ό,τι ο μέσος όρος, έχουν ένα στρατηγικό συμφέρον να ανοίξουν και οι υπόλοιποι και αυτό ισχύει και για τους Ευρωπαίους. Υπάρχει μια στρατηγική ε, τοποθέτηση η οποία θα πρέπει να αποδώσει. Αλλά και γι' αυτό θα χρειαστεί οι Αμερικάνοι να ε, καλύψουν ε, και να έχουν πλειοψηφία στο Κογκρέσο, πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές. Όσον αφορά τη γεωργία, η συζήτηση στον ΠΟΕ ε, μοιάζει με τις συζητήσεις που έχετε μεταξύ Ευρωπαίων Δηλαδή η γεωργία είναι όπως ε, τα, οι κάλτσες και τα ελαστικά. Πρέπει να ανοίξουμε την αγορά, να βοηθήσουμε τον καταναλωτή, θα είναι προς όφελος όλων, άρα η γεωργία πρέπει να προσωμιαστεί στις άλλες, ε, στους άλλους τομείς. Άλλοι πάλι λένε δεν είναι το ίδιο. Καταρχήν ε, διότι δεν έχει κανείς την ίδια σχέση με τη γεωργία που έχει με τα παπούτσια του, διότι υπάρχουν ιδιομορφίες και μας το εξηγούν. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και κλιματολογική και περιβαλλοντολογική. Εν ολίγης υπάρχουν και οι δύο παρατάξεις, όπως υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και η συζήτηση αυτή δεν πρόκειται να επιληθεί με ε, τον κύκλο της Ντόχα. Δηλαδή δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα θέματα θα λυθούν σαν τις κάλτσες. Θα πρέπει βάσει των ε, τωρινών διατάξεων